Έχουμε οικονομολόγους και ε, ειδικού σε θέματα χρηματοπιστωτικών γυναίκες πολύ καλές και στις επιχειρήσεις και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στις τράπεζες. Υπάρχει ποικιλία και ισορροπία εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια και η διαδικασία λήψεων, α, αποφάσεων όταν ε, υπάρχει αυτή η μεγαλύτερη ισορροπία είναι και πιο ισορροπημένη και αυτή. Οι άνδρες ε, πολλές φορές παίρνουν αποφάσεις πιο ρηψοκίνδυνες ε, ε, με λιγότερη ίσως υπευθυνότητα. Δεν το λέω αυτό, το βλέπουμε και το συνάγουμε από δεδομένα που έχουμε συλλέξει από πολλούς ε, ε, από πολλούς φορείς. Οπότε καλό είναι να υπάρχει αυτή η ισορροπημένη εκπροσώπηση για να είναι και η ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Αν λοιπόν να εργαστούμε καλύτερα στο μέλλον ε, επί των διαδικασιών που θα εγγυηθούν καλύτερη ισορροπία των διαφύλων, αυτό θα οδηγήσει και σε καλύτερο ανταγωνισμό και στην οδηγία για την εκπροσώπηση των γυναικών ε, στα ΔΣ. Το πρώτο βήμα είναι η εμπειρία, η ποιότητα, η επαγγελματική ικανότητα. Και μετά, δεύτερο κριτήριο, το υποεκπροσωπούμενο φύλλο. Νομίζω είναι δίκαια αυτά τα κριτήρια και ουσιαστικά είναι ουδέτερο προς το φύλλο, γιατί μπορεί την προτεραιότητα μία μέρα να την έχει ένα άνδρας. Άρα νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνουμε πιο δίκες αυτές τις διαδικασίες. Ως ε, αρμόδια ε, για θέματα ισότητας ε, είμαι, έχω τα, ασκώ τα καθηκοντά μου εδώ και πέντε χρόνια. Άκουσα κάποιον να λέει ότι είμαστε διαφορετικοί άνδρες από τις γυναίκες. Φυσικά είμαστε διαφορετικοί, σκεφτόμαστε διαφορετικά, γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει ισορροπημένη εκπροσώπηση. Είμαστε διαφορετικοί όλοι ω άτομα. Εγώ έρχομαι από μια πολιταρχική χώρα, αλλά ε, όταν ακούω ε, για ισότητα, κάπως έτσι... Ε, γίνομαι νευρική γιατί είμαι από μια χώρα που επέβαλε ε, την ισότητα. Λοιπόν, ε, δεύτερος μύθος, ποσοστώσεις για την οδηγία στις, για τις γυναίκες στα που θέλετε να χρησιμοποιηθεί και για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. σαν ε, να λέγεται από κάποιους ότι με τις ποσοστώσεις ε, ένας φανταστικός ε, άνδρας με καταπληκτικά προσόντα θα την από μια γυναίκα. Όχι, αυτό δεν αληθεύει. Μιλάμε για δίκαιο ανταγωνισμό. Εγώ αυτό προωθώ. Πρέπει να δούμε τι έγινε, να διδαχθούμε από τις ανεύθυνες αποφάσεις, τις αποφάσεις και την κρίση δεν ήταν Lehman Sisters η τράπεζα, αλλά ήταν Lehman Brothers. Ίσως γι' αυτό να ήταν έτσι κατάσταση. Επίσης βλέπω και πολλούς νέους ανθρώπους όταν ε, έρχομαι σε επαφή με νεαρές γυναίκες, ε, ε, φοιτήτες κτλ. Οι γυναίκες δεν μιλάνε τόσο για τις διακρίσεις. Θέλω να προχωρήσουν. Και πρέπει να τις βοηθήσουμε τις γυναίκες να προχωρήσουν, να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να ε, είναι έτοιμες να αναλάβουν υψηλά αξιώματα. Γιατί χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση με βάση πολλές έρευνες είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για τις γυναίκες. Γι' αυτό δεν διεκδικούν ένα υψηλό αξίωμα. κάπως αποφεύγουν ε, να, να εκτέθουν σε κάποιο κίνδυνο για τον κύριο Σόσνη. φυσικά και δεν συμφωνώ με αυτά όσα είπε. Ήμουν εδώ χθε, κυρίε και κύριοι, και συζητήσαμε την υδατοκαλλιέργεια, την προστασία των ζώων και των ψαριών. Άκουσα χθε ότι τα ψάρια δεν χρειάζονται την προστασία μας, δεν αξίζουν την προστασία μας, γιατί δεν ψηφίζουν και δεν πληρώνουν φόρου. Άρα πιο ήπια ίσως ήταν η γλώσσα που άκουσα σήμερα. Ευχαριστώ για τις γυναίκες εννοώ. Και ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιούροβα. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, ε, η κυρία Τσιώτη για μια ακόμη φορά έχει το Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αν και τα κλείδι θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι όσον αφορά τους διορισμούς στα όργανα του νομισματικού και οικονομικού τομέα το Συμβούλιο είναι ταγμένο στην πρόθεση της ισότητας θα δρά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ελπίζω επίσης ότι μπόρεσα να διευκρινίσω τον ρόλο του Συμβουλίου στις σχετικές διαδικασίες επιλογής. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Τσότ. Πέντε προτάσεις ψηφίσματος έχουν κατατεθεί. Εδώ ολοκληρώνω τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Πέμπτη. Πρέπει να κάνουμε σύντομο διάλειμμα. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φίλοι μου, είναι σημαντικό για μας να μπορούμε να συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πελεγκρίνη, το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται στο κέντρο της δημοκρατίας. Είναι η καρδιά της. Και μετά την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γαλλικής Δημοκρατίας. Θέλουμε να ξέρουμε όλα τα κράτη-μέλη πώς τοποθετούνται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση αυτή είναι εντελώς ανοιχτή ως διαδικασία για το μέλλον το σημαντικότερο είναι να ενισχύσουμε για μας τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου ως προς το θέμα της μετανάστευσης. Αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει ως πρώτο μέλημα. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την ε, μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου και ζητούμε να λάβει σχετική απόφαση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όμως ταυτόχρονα θέλουμε να κάνουμε πιο πολλή δουλειά στην Αφρική. Θέλουμε να επενδυθεί χρήμα στην Αφρική είναι σημαντικό. Ε, είναι επίση σημαντικό να προσέξουμε τις ε, κοινωνικές μας πολιτικές. Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίζει το μέγεθος της ανεργίας των νέων ως φαινομένου. Ε, είναι κάτι που επηρεάζει το τι συμβαίνει και στην πραγματική οικονομία, που και αυτή πρέπει να ενισχύσουμε, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα καταπολεμήσουμε τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Είναι σημαντικά όλα αυτά για το Ευρωκοινοβούλιο. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι σημαντικό να το δούμε και υπό το φως του τι ψηφίσαμε προσφάτως για την Κίνα. Η κινέζικη πολιτική και, για, και αυτό για μας είναι προτεραιότητα. Και υπάρχουν και άλλα σημαντικά στην ε, ατζέντα μας πριν τις εκλογές. Το Brexit Πολύ σημαντικό. Ήταν εδώ χθε η κυρία Μέη. Αλλά και γι' αυτό και για όλα τα άλλα θέματα ήταν σημαντικό να ξέρουμε τη θέση της Σλοβακίας. Σας ευχαριστώ. Vi prego di registrarvi per eh, il Σας παρακαλώ να καταγραφείτε για τη διαδικασία Catch the Eye. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να συμμετάσχω στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Αποτελεί τιμή και προνόμιο για μένα να είμαι εδώ σήμερα στον οίκο της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Η ιστορία του ανθρώπου είναι η ιστορία της δημιουργία ιδεών για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό σηματοδοτήθηκε και από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από 60 χρόνια. Αυτό δρομολόγησε τις ε, δημοκρατικές αλλαγές στην Τσεχοσλοβακία πριν από 30 χρόνια. Εργαζόμεθα για την ειρήνη, την ευμερία και την πρόοδο στην Ευρώπη. Και όλα αυτά έφεραν και σε εμά σταθερότητα, ελευθερία και όντω ευημερία. Έφεραν επιτυχία ακόμα και σε μικρές χώρες όπως η Σλοβακία εν προκειμένου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ιστορία ξανάρχισε για εμάς το 1989 λόγω τη επιθυμία μας για ελευθερία, για δικαιώματα του ανθρώπου, για τεχνολογική πρόοδο. Γίναμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση και του ΝΑΤΟ πριν από 15 χρόνια και ανήκουμε πλέον εκεί που ανέκαθεν ανήκουμε στο ευρωπαϊκό και βορειοατλαντικό σύστημα αξιών. Η ιστορία της Σλοβακίας από τότε είναι μια ιστορία επιτυχιών. Παρ' όλα αυτά ο δρόμος δεν ήταν πάντοτε εύκολος. Περάσαμε από οικονομικές δυσκολίες, από τις δυσκολίες της μετάβασης, αντιμετωπίσαμε υψηλή ενέργεια, ανεργία, αναδημορφώσαμε την οικονομία μας, δημιουργήσαμε δημοκρατικούς θεσμούς στο νέο κυρίαρχο κράτος. Άφησαμε πίσω μας την κρίση και αντεπεξήλθαμε στις προκλήσεις της συνταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέλλον και στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά ήταν μια διαδικασία με όλους κερδισμένους. Είχαμε την ευκαιρία να εξυγχρονιστούμε, να πάμε μπροστά. Όλα τα κράτη-μέλη έγιναν πλέον πιο σταθερά μέσα στην ενιαία αγορά. Σήμερα η Σλοβακία είναι πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Είμαστε μεταξύ των χωρών μελών με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Είμαστε μέλη της Ευρωζώνης, έχουμε χαμηλή ενεργεία και από χώρα αποχωρούν των μεταναστών. Είμαστε μια χώρα της οποίας ο πληθυσμός αυξάνεται. Το κλίμα άλλαξε και αυτό στη χώρα μου. Οι πολίτες μας απολάβουν ελευθερία, και έχουν γίνει μάλιστα και πιο απαιτητικοί όσον αφορά του πολιτικού του εκπροσώπους. Αξιοποιούμε λοιπόν αυτέ τι προοπτικέ, συνεχίζουμε να εξυγχρονίζουμε τη χώρα μα, την κοινωνία των πολιτών. Είμαστε μια χώρα στην οποία τα μέσα είναι ελεύθερα. Βεβαίω, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα σε πολλού τομεί, ιδιαίτερα στον τομέα τη εκπαίδευση, τη έρευνα, τη καινοτομία. Εκεί υπάρχουν πολλέ δυνατότητες, τον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης, την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αποτελέσουμε έμπνευση και για άλλες χώρες. Και ξέρουμε ότι όπου υπάρχει θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ο Στεφάνι Μεγάλος διπλωμάτης και ιδρυτής της Σλοβακίας το 1918 είπε ότι αν θέλουμε δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να επιτύχουμε. Μετά από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό συνέχισε να ισχύει. Όπως προείπα, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες για την ένταξή μας στο Σέγγεν, στην Ευρωζώνη, αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ να προσπαθούμε. Διότι ανέκαθεν πιστεύαμε στα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το φυσικό μας περιβάλλον. Εκεί ανήκουμε. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση. Κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας στείλαμε το ίδιο ακριβώς σαφές μήνυμα. Ένα μήνυμα ενότητας λίγο μετά από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Βρετανία. Συνεχίζουμε λοιπόν, όμως δεν είμαστε στο απειρόβλητο. Υπάρχει δυνατότητα πρόοδου στον τομέα της ελευθερίας των μέσων. Γνωρίζουμε τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και το ζήσαμε και στην Σλοβακία. Αυτό όμως είναι και ένδειξη, αν όχι απόδειξη, της οριμότητας της δημοκρατίας μας. Μετά από την ε, δολοφονία του Κούτσιακ και της ε, φίλη του λάβαμε μέτρα εντό λίγων εβδομάδων. Δολοφονήθηκαν δύο νέοι άνθρωποι και αυτό αποτέλεσε ένα τεράστιο κλονισμό για όλη την κοινωνία της Σλοβακίας. Ο στόχο ήταν ένας και μοναδικός. Να εντοπίσουμε, να εντοπίσουμε και να τιμωρήσουμε τους δολοφόνους. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δει στην ομάδα παρακολουθήσης του κρατούς δικαίου για τη βοήθεια και την συνεργασία που μας εξασφάλισαν ως σήμερα. Δεχθήκαμε επικρίσεις κατά καιρού, είναι αλήθεια, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και την Europol για τη βοήθειά της να προσαγάγουμε τους πρώτους υπόπτους οι οποίοι τώρα είναι υπόδικοι. Σήμερα, εκ μέρους του σλοβακικού λαού, θέλω να επιβεβαιώσω ότι αυτές οι δύσκολες μέρες αποτελούν παρελθόν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα για το μέλλον, να ερχόμαστε πιο κοντά στις άλλες χώρες και να υλοποιούμε τις ευθύνες που μας αναλογούν για να διαμορφώσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Σε λίγο έχουμε προεδρικές εκλογές και είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες μας θα αποδείξουν την οριμότητά τους επιλέγοντας υποψηφίους ε, υπέρ της Ευρώπης υπέρ του Ευρωπαϊκού Ιδεώδους. Το κόμμα που εκπροσωπώ, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα που κυβερνά, δεν θα μπορούσε να έχει άλλο υποψήφιο εκτό από τον κύριο Σεφκοβίτς, τον σημερινό αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Δεν υπάρχει άλλος πιο ε, υπέρ της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, οι επιτυχίες της Σλοβακίας σε κάποιο βαθμό εξηγούνται από την ιστορία μας. Η κεντρική Ευρώπη είναι ο φυσικός μας χώρος. Εκεί είναι η ιστορία μας, η γεωγραφία, ο πολιτισμός μας. Εν τέλει, η περιφερειακή συνεργασία είναι και η πεμπτουσία της επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γαλλογερμανική συνεργασία, η Βαϊμάρη, το Μπενελούξ, η Βαλτική, ακόμα και η ομάδα είναι πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν με ιδέες και ενισχύουν την Ένωση. Η Σλοβακία αυτή τη στιγμή προεδρεύει τη ομάδα Βίσεγκρατ. Ο βασικό μα στόχο είναι η θεματική μα να είναι μια θετική και υπέρ τη ευρωπαϊκή περαιτερωνοποίηση. Φυσικά υπάρχουν διαφορέ απόψεων, υπάρχουν επικρίσει αριστερά και δεξιά, υπάρχουν παρανοήσει, όμω σε αυτού του δύσκολου καιρού οφείλουμε όλοι να συνεχίσουμε να προσπαθούμε γύρω από το ίδιο τραπέζι Οφείλουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να επιλύουμε τις διαφορές μας μέσω διαλόγου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το απότοκο ενός ισχυρού οράματος και των προσπαθειών πολλών γενεών. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε τώρα, ειδικά τώρα που αντιμετωπίζουμε δραματικές εξελίξεις. Έχουμε προκλήσεις ε, πανταχώθεν από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό, από το περιβάλλον μας. Βλέπουμε τις φιλοδοξίες της Κίνας, της Ρωσίας και αυτό ζητά από εμά μια ενιαία απάντηση. Βλέπουμε την μεταβολή του κλίματος που επιφέρει απροσδόκητες επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Είμαστε μάρτυρες τεχνολογικής πρόοδου. Εμείς θα επιζήσουμε ως Ευρώπη αν παραμείνουμε στο προπήριο των τεχνολογικών αλλαγών και της καινοτομία. Για να το πετύχουμε αυτό, οι κυβερνήσεις μας πρέπει να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. Έχουμε αυξανόμενες, ενδυνόμενες κοινωνικές ανισότητες. Βλέπουμε να καταραίει το κοινωνικό συμβόλαιο. Έχουμε να κάνουμε με την γύρανση του πληθυσμού. Έχουμε να κάνουμε με διαφορές περιφερειακές ε, ή μεταξύ χωρών, κάτι το οποίο δεν ε, συνεισφέρει στο αίσθημα της ενότητας. Πολλοί πολίτες μας αισθάνονται ότι έχουν μείνει πίσω, ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και αυτό ε, συνδυάζεται με την μαζική μετανάστευση από τρίτες χώρες, κάτι το οποίο επιτείνει την κρίση στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για την δημοκρατία, για τους ανθρώπους, για το σχέδιό μας, για το μέλλον. Όταν οι άνθρωποι, όταν οι πολίτε μα δεν βρίσκουν απαντήσει σε εμά, θα κοιτάξουν αλλού. Η έλλειψη επικοινωνία μπορεί να είναι και το εκολαπτήριο για τις ψευδοειδήσει. Ένα παράδειγμα αυτού του αποτελέσματο, ένα τέτοιο απότοκο είναι και το βρετανικό δημοψήφισμα. Ο απομονωτισμός, ο προστατευτισμός και ο εθνικισμός δεν αποτελούν λύση. Η δική μας απάντηση δεν είναι ο κατατεμαχισμός, ο κατακαιρματισμός, ο περικλεισμός στα εθνικά μας κράτη. Είναι η περισσότερη ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιας δύναμης. Κυρίες και κύριοι, όπως έκανε και οι 17 συναδελφοί μου, θα έχω και εγώ το θάρρος να καταθέσω το δικό μας όραμα για το μέλλον. Ένα όραμα μιας Ένωση ελκυστική για του πολίτε, που μπορούν να εμπιστευθούν οι πολίτε, την οποία θέλουν να υποστηρίξουν. Αυτό παραμένει το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πρατισλάβα. Θέλουμε πρώτα απ' όλα μια ένωση ενωμένη, ευημερούσα, που παρέχει ασφάλεια. Δεύτερον, μια ένωση η οποία διαδραματίζει παγκόσμιο ρόλο. Ένα ρόλο στα παγκόσμια πράγματα ένα, μια ένωση η οποία είναι ειλικρινής προς τους πολίτες της και τους φροντίζει και η οποία κάνει για το μέλλον της ό,τι περνάει από το χέρι της. Χρειάζεται ένας κοινό δρόμος για να υλοποιήσουμε βεβαίως αυτό το όραμα. Το δικό μου ερώτημα είναι πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά. Πρώτον, χρειάζεται να παραμείνουμε ενωμένοι. Η ενότητα ήταν η λέξη που χρησιμοποίησαν τις περισσότερες φορές οι συνάδελφοί μου που απευθύνθηκαν σε αυτό το κοινοβούλιο και πιστεύω ότι έχουν δίκιο. Χωρίς ενότητα θα υποταχθούμε απλούστατα στις αποφάσεις άλλων τρίτων. Δεν θα είμαστε αξιόπιστοι στην προσπάθεια εάν δεν υπερπηδήσουμε τα τελευταία υπολείμματα της διαχωριστικής γραμμής Ανατολής Δύσης. Να αφήσουμε πίσω μας τα στερεότυπα τα οποία απλώς υπενθυμίζουν τις διαφορές μας. Σας θυμίζω τον Μίλεν Χότζα ο οποίος ήταν πρόεδρος, ε, πρωθυπουργός, ε, με συγχωρείτε, της Τσεχοσλοβακίας, την περίοδο Το 42 ε, έγραφε «Η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν αφορά μόνο τη Δύση, δεν θα κατασκευαστεί εκεί, χρειάζεται και την κεντρική Ευρώπη. Και τα κοινά δημοκρατικά ιδεώδη χρειάζονται και αυτά για να έχουμε ελπίδα για το μέλλον. Πιστεύω προσωπικά ότι πέραν των διαφορών και των συνόρων έχουμε ένα κοινό συμφέρον. Πρέπει να επικοινωνήσουμε, πρέπει να κατανοήσουμε ένα τον άλλον και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, εκατέρωθεν, ένθεν, κακήθεν. Πρέπει να υπερπηδήσουμε τα παλιά εμπόδια, τις παλιές διαφορές και για να αναφέρω δύο παραδείγματα, η απόσπαση εργαζομένων ή τα πρότυπα για τα τρόφιμα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα στο οποίο αποτύχαμε να επικοινωνήσουμε. Μιλώ για την μετανάστευση. Εκεί πρέπει να βρούμε μία λύση η οποία θα αποδίδει και για τους μεν και για τους δε. Η μετανάστευση πρέπει να τύχει κανείς διαχείρισης. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει εν τέλει να υπηρετεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η πολιτική ενότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την οικονομική σύγκληση και συνοχή. Με άλλα λόγια, η ευημερία πρέπει να υπηρετήσει το κοινό καλό. Πρέπει να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση και να πατάξουμε την φοροαποφυγή από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει οι φόροι να καταβάλλονται στις χώρες ακριβώς εκεί που γεννάται ο πλούτος. Πρέπει να πατάξουμε επίσης τις εντυνόμενες διαφορές και ανισότητες της κοινωνίας μας. Ο πλούτος πρέπει να διανεμηθεί με τρόπο ισότιμο εισαγωγή ενό ελάχιστου ευρωπαϊκού μισθού νομίζω ότι θα είναι ένα τρόπο επίδειξη ελεγγύης. Η κυβέρνησή μου είναι ενταγμένη στην υποστήριξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα. Είναι υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων, είναι η κοινωνική διάσταση του μέλλοντος της Ευρώπης. Η Σλοβακία είναι επίσης υπέρ της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων. Αυτό ακριβώς θα επιτρέψει σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις να δράξουν τις ευκαιρίες τη ενιαία αγορά. Θέλω να εκφράσω λοιπόν την ικανοποίησή μου για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία. Έχουμε την φιλοδοξία να την φιλοξενήσουμε στην πρωτεύουσά μα. Δεύτερον, πρέπει, όπω είπα, να διαδραματίσουμε έναν ρόλο στα παγκόσμια δρόμενα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει ρόλο παγκόσμια διάσταση. Αυτό είναι ο ρόλο μα, αυτή είναι η θέση μα. Πρέπει να ενώσουμε τι προσπάθειέ μα, να ενώσουμε τι δυνάμει μα και στον τομέα τη άμυνα. Η Σλοβακία είναι σαφώς υπέρ της μόνιμης διαρθρωμένης, δομημένης εργασίας στο πλαίσιο της Άμυνα και της ασφάλειας, στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΟ, διασφαλίζοντας συμπληρωματικότητα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Έλεγα λοιπόν παγκόσμιος ρόλος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελοπίσουμε και τις δεσμεύσεις μας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Δεν είμαστε απομονωμένοι, είμαστε ανοιχτοί, είμαστε ανοιχτοί σε όλους όσους πληρούν τα κριτήρια ακόμη και σε αυτούς που κάποτε έφυγαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο στρατηγικός μας ρόλος. Αν δεν το πράξουμε εμείς, κάποιος θα τρέξει να πληρώσει το κενό. Και ταυτόχρονα, παγκόσμιος ρόλος σημαίνει να είμαστε μια σπουδαία οικονομική δύναμη, να έχουμε ένα ισχυρό νόμισμα, Βασισμένοι σε έναν παγκόσμιο ρόλο και στον τομέα του εμπορίου. Πρέπει να παραμείνουμε στο προπύριο σαν αφορά τις θέσεις αυτές. Τρίτον, πρέπει να είμαστε έντιμοι έναντι των συμπολιτών μας. Δεν μπορούμε να υποσχόμαστε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι θα χρειαστεί σκληρή δουλειά. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Οι πολίτες μας χρειάζονται ένα σαφές όραμα, ένα όραμα το οποίο όμως μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πράξεις τους πολίτες μας και κυρίως τους νέους πολίτες μας. Πρέπει να τους κάνουμε συμμετόχους στο όραμα αυτό. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ενστερνιστούν το όραμά μας. Να δώσουμε ένα τέλος στην εντύπωση που δίνουν οι Βρυξέλλες, ότι είναι μακρινές. Ας αφήσουμε πίσω λοιπόν αυτούς που λένε το αντίθετο αλλά ας αντιταχθούμε με επιχειρήματα, όχι περιγελώντας τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισχυρή κοινότητα. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η συλλογική μας ταυτότητα. Ξέρετε, το θέμα είναι και η προσωπική εμπλοκή του καθενός, χωρίς να αφήνουμε πίσω μας την εθνική μας ταυτότητα. Ενότητα είναι ενότητα αξιών, ενωμένη στην πολυμορφία, με τα δικά μας εθνικά, περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά. Τέλος, κάτι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον επιτέλους. Σύντομα, έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές. Εσείς, οι πολιτικές ομάδες, οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, θα έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε το δικό σας ρεαλιστικό όραμα για την Ευρώπη. Ο διάλογος για την Ευρώπη θα είναι έντονο σε πολλά επίπεδα, σε πολιτικό επίπεδο, στο επίπεδο των πολιτών, στο εθνικό επίπεδο και το περιφερειακό επίπεδο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίο ε, δρομολόγησε μια ζωντανή συζήτηση, ένα διάλογο για το μέλλον τη Ευρώπη και συμφωνώ με τι θέσει του πρόεδρου Μακρόν. Δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε στο σύνδρομο της παρέτησης. Όχι, χρειαζόμαστε μια ζωντανή ένωση και να σε εμά, του ηγέτε, να βρούμε τον κοινό δρόμο με μηχανισμού οι οποίοι εμπνέουν εμπιστοσύνη στου πολίτε. Χρειαζόμαστε ελευθερία, πρόοδο και προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αποστελέσουμε τις τέσσερις ελευθερίες που βρίσκονται, που αποτελούν την πεμπτουσία της ενοποίησης. Χρειαζόμαστε μια ένωση και έναν διάλογο περί στρατηγικής. Τι προσδοκούμε ως τα μέσα του 21ου αιώνα. Θα χρειαστεί να αναδιαμορφώσουμε την Ένωση το κλίμα, την οικονομία. Χρειαζόμαστε μια μετάβαση η οποία θα είναι δίκαιη κοινωνικά για τους πολίτες, δίκαιη για τις επιχειρήσεις μας. Ένα σημαντικό θέμα για το μέλλον της οικονομίας μας είναι η ψηφιοποίηση και η αυτομετοποίηση. Βεβαίως υπάρχουν ανησυχίες ότι ο κόσμος δεν θα έχει αρκετές δουλειές λόγω των ρομπότ, λόγω της αυτομετοποίησης. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και ανησυχίες για την έλλειψη εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα. Είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούμε περισσότερου τέτοιου εργαζομένου στο προσχέ μέλλον. Και τρανή απόδειξη αυτού είναι ότι οι χώρε με τα περισσότερα ρομπότ, η Γερμανία, η Νότιο Κορέα, η Σιγκαπούρη, έχουν τους χαμη... τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 150 ρομπότ για κάθε 10.000 θέσει εργασία στη Σλοβακία. Αυτό είναι πάνω από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές φορές πάνω από τον μέσο όρο της κεντρικής Ευρώπης. Λοιπόν, ας μην φοβηθούμε την τεχνολογική πρόοδο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσαρμοστούμε με τρόπο ευφυή. Χρειαζόμαστε ευφυείς πολιτικές. Και αν με ρωτήσετε πώς βλέπω το μέλλον. Ναι, χρειαζόμαστε τα σωστά εργαλεία για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο τρέχον προπολογισμό της Ένωσης είναι μόνο το 1% του συνολικού ΑΕΠ. Λοιπόν, ας μην ξεχνούμε και την συνοχή και τη σύγκληση στο πλαίσιο του επομένου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, να μην ξεχάσουμε λοιπόν και τη συνοχή. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι θα γίνει με τι απομακρυσμένε και τι φτωχότερε περιοχέ για να μπορέσουν και αυτέ να συμβάλλουν στην οικονομική μα ε, ανάπτυξη, ακόμα και σε αντίξωε οικονομικέ συνθήκε και δύσκολου καιρού. Ε, προανέφερα ότι πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον μας Παρακαλώ. Πώς να μιλήσουμε για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο χωρίς να έχουμε ένα ξεκάθαρο και σαφές μακρόπνο όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η προσέγγιση. Πρώτα, να δούμε τι μπορεί να έχουμε στο επίπεδο του προπολογισμού και μετά να αποφασίσουμε τι θα πληρώνει, τι θα καλύπτει αυτός ο προπολογισμό. Αλλά δεν είναι αυτό η καλύτερη επιλογή. Πρώτα πρέπει να δούμε τι θα γίνει τα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια, ποιε είναι οι προτεραιότητέ μα και μετά να αποφασίσουμε τι είδου προπολογισμό χρειαζόμαστε. Αυτή την προσέγγιση την προτιμάω εγώ από αυτό που κάνουμε τώρα. Και για τις νέες τεχνολογίες. Ας το πούμε ξεκάθαρα και δεν μιλώ εδώ για το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά γενικώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορούμε να προλάβουμε τις εξελίξεις στον κλάδο αυτό. Διαρκώς ε, είμαστε πίσω. Ε, υπάρχει τεχνολογική επανάσταση γύρω μας, αλλά δεν βλέπουμε καμιά επανάσταση στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Διαρκώς καθυστερούμε. Ε, ήδη προσπαθούμε να ρυθμίσουμε κάτι που χρησιμοποιεί ο κόσμος ήδη στην πράξη. Και προβλέπουμε τέτοιε ρυθμίσει που τελικά είναι υπέρμετρε, υπερβολικέ και καταπνίγουν. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τη ΗΠΑ, τι χώρε τη Νοτιοανατολική Ασία και γιατί αλλού ε, ευνοείται η ανάπτυξη αυτού του κλάδου με τόσους πολλούς κανονισμούς που έχουμε, δεκάδες. Γι' αυτό λοιπόν ας σκεφτούμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να είναι ευέλικτο, να μην κοιτάζουμε να διαβεβαιώσουμε την κάθε παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής μας. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε έτσι την ψηφιακή επανάσταση. Κάτι βασικό χρειαζόμαστε σε ένα πλαίσιο που να ε, δίνει κάποιες ε, αδρές γραμμές, αλλά εμείς ως πολιτικοί πρέπει να δρούμε και με ταχύτητα. Εάν μιλάμε για την τεχνολογία 4.0, ε, πρέπει να φροντίσουμε και οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί μας να είναι στο επίπεδο του 4.0. Διότι για την ώρα είμαστε κάπου κοντά στο 3.0, αλλά το 4.0 δεν το έχουμε πετύχει ακόμα πουθενά στο επίπεδο των κυβερνήσεων. Κυρίες και κύριοι, οι ευρωπαϊκές εκλογές πλησιάζουν βήματα χ. Πρέπει και εμεί λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε με ταχύτητα για να αντιμετωπίσουμε τι ε, ψευδεί ειδήσει, τι κυβερνοαπειλέ και την προπαγάνδα. Πρέπει να μιλήσουμε στον κόσμο για τη σημασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για το πόσο σημαντικό είναι να ψηφίσουν για την καθημερινότητά του, ε, να καταλάβουν ότι εκλογέ έχουν σημασία. Είναι μόνη του ευκαιρία να αναλάβουν εκείνη το πιδάλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην αποφασίσουν άλλοι στη θέση του. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας και να ολοκληρώσω την ομιλία μου με τα εξή λόγια Ενό από τους ιδρυτέ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ναι. Ο κόσμος δέχεται την αλλαγή μόνο όταν πιέζεται από την ανάγκη και αναγνωρίζει την ανάγκη μόνο όταν η κρίση πιέζει τον ίδιο. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε διαρκώς. Πρέπει να φέρουμε αλλαγέ και να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ελκυστική για όλου. Μια ένωση που να είναι σε θέση να διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος και να προετοιμαστεί για να ε, καλπάσει στο μέλλον. Χρειαζόμαστε ένα όραμα. Μια ελκυστική ένωση που να μπορούν να εμπιστευτούν οι πολίτε και να τη στηρίξουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρωθυπουργέ για την ε, ομιλία σας. Επόμενος ε, ε, για να πάρει το λόγο είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ. Μποντζόρνο κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Πέτερ, θα σας θα μοιραστώ μαζί σας ένα μυστικό. Δεν κοιμήθηκα και πολύ λόγω της κυρίας Μέη απόψε το βράδυ αλλά παρόλα αυτά κοιμήθηκα γιατί ονειρεύτηκα τη Σλοβακία και την Πρατισλάβα. Διότι χθε διαπραγματευόμενος ε, με την κυρία Μέη σκέφτηκα την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη της Μπρατισλάβα του Δεκεμβρίου του 2016, τρεις μήνες μετά την απόφαση των Βρετανών να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνησή σας, ήσασταν μέλος της κυβέρνησης ε, και τότε, και σε ό,τι αφορά την Σλοβακή Προεδρία και τον απολογισμό της ε, έχετε καταφέρει πολλά, δέχτηκα για πρώτη φορά στην ιστορία να φιλοξενήσει ε, σύνοδο κορυφής ε, των 27, διότι η Σλοβακική κυβέρνηση θεωρούσε ότι το Brexit είναι το παρελθόν και εμείς πρέπει να προετοιμάσουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι πιστεύαμε και εμείς και αυτό έγινε και στην Πρατισλάβα. όπου έμεινε και η έκφραση του οδικού χάρτη της Μπρατισλάβα. Λίγες ημέρες μετά ε, την ομιλία μου για την κατάσταση της Ένωσης ε, εδώ, για πρώτη και ίσως και τελευταία φορά, 27 πρωθυπουργοί χαιρέτησαν το περιεχόμενο της ομιλίας, κάτι που ποτέ δεν είχε ξανασυμβεί και δεν θα ξανασυμβεί και ποτέ. Όμως ε, το έχω συγκρατήσει στο μυαλό μου ε, αυτή τη διάσκεψη κορυφής Βαρσιλάβα ω μια ξεχωριστή στιγμή γιατί ήταν ε, μια στιγμή όπου με αποφασιστικότητα και θάρρος έστω και μικρά βήματα προχωρήσαμε εκείνο το βράδυ μαζί με τη Βρετανική κυβέρνηση για τις προϋποθέσεις και τους όρους καθώς και τις ε, συνέπειες του Brexit. Χθες το βράδυ, τα πω τη νύχτα, είπα ότι αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία, αλλά τρίτη δεν θα υπάρξει. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων να στηρίξουν αυτή τη βρετανική και ενωσιακή προσέγγιση υπό τη μορφή του συμπεφωνημένου αυτού κειμένου για να έχουμε συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέτερ, θέλω να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη που συνεχώς μας παρέχει η Σλοβακική κυβέρνηση. Και θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στις προσπάθειες της Σλοβακίας για την τροποποίηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τη δημιουργία της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής για την εργασία. Και η κυβέρνηση, η χώρα ε, που θέλει να φιλοξενήσει, μάλλον ε, ο αριθμό των χωρών που έχουν εκφράσει τη βούλησή του να φιλοξενήσουν αυτή την αρχή είναι πολύ περισσότερε από αυτέ που ήθελαν να φιλοξενήσουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Χαίρομαι που σα άκουσα να λέτε ότι σας αρέσει ο κοινωνικός πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο περισσότεροι πρωθυπουργοί το λένε αυτό, όχι μόνο εδώ, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όχι μόνο εδώ, αλλά και σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών, τόσο λιγότερο απομονωμένο νιώθω εγώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σλοβακική κυβέρνηση μα βοήθησε τα μάλα ώστε να ε, υλοποιήσουμε το κοινωνικό πυλώνα στο Γκέτεμπορκ όπου και το λέω για αυτούς που συνεχώς ε, το διεκδικούν περιλαμβάνεται η ανάγκη παντού στην Ευρώπη να καθιερωθεί ένας ελάχιστος, ένας κατώτατο μισθός. Δεν είναι κάτι που πρέπει στι τελευταίες εβδομάδες, είναι μια ιδέα που την έχουμε εκφράσει από τότε που εμείς αναλάβαμε καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω το στόματερο δυνατόν ε, να γίνει πραγματικότητα. Το ίδιο ισχύει και για ένα ελάχιστο εισόδημα ε, για όλες τις χώρες της Ένωσης. Μιλήσατε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και είπατε πολύ σωστά ότι πρώτα πρέπει να συμφωνήσουμε για τις πολιτικές και εν συνεχεία για τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών των πολιτικών. Ακριβώς έκανε αυτό το πράγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή ακριβώς την προσέγγιση ακολουθήσαμε. Και αυτό ανταποκρίνεται και στις ε, επιθυμίες που εκφράστηκε. Είπατε και εσείς δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε την ανάγκη που υπάρχει. Πρέπει να παραμείνουν οι πολιτικές συνοχής. Εγώ είμαι μεγάλος υπέρμαχος και λάτρης ε, της πολιτικής συνοχής. Βέβαια, έπρεπε να λάβουμε ταυτόχρονα υπόψη και πρέπει να το είπατε κι εσείς, ε, πρέπει να προωθήσουμε πολιτικές καινοτομίας, εξυγχρονισμού, ψηφιακές πολιτικές στην Ευρώπη της Άμυνας. Όλα, τα, όλα αυτά τα κάναμε. Και αν δεν είχαμε επανεξετάσει την ε, πολιτική και την ε, ευρωπαϊκή κοινή γεωργική πολιτική, θα είχαμε φτάσει σε 1,48% του ΑΕΠΑ. 1,41. Αλλά αυτό δεν θα γινόταν δεκτό ποτέ, οπότε έπρεπε να κάνουμε επιλογές. Όπερ και επράξαμε. Η Σλοβακία ασκεί την προεδρία του Βίζεγκρατ. Και θέλω να δράξετε αυτή την εμπειρία, ώστε αυτή η συζήτηση, η αχρίαστη συζήτηση που έχουμε μεταξύ των Ανατολικό Κέντρο Ευρωπαίων και των Δυτικοευρωπαίων να πάψει. Θα πρέπει ε, η Ευρώπη να αναπνέει και με τα δυο της πνευμόνια. Άρα πρέπει να κάνουμε πάντα δυνατό ώστε να μην ε, σφιχτεί ούτε το ένα ούτε το άλλο μέσα στο ίδιο σώμα. Όλοι μας ε, έχουμε τη συμβολή μας. Και δεν είναι μόνο η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, κάποιες κυβερνήσεις της Ανατολικής Ευρώπης που είναι υπεύθυνε για τη γελία ενίοτε αυτή η αντιπαράθεση που σίγουρα είναι επιζήμια και ελπίζω να εκμεταλλευτείτε το γεγονό ότι προεδρεύετε και ε, του Βίσεμπραντ αυτή την περίοδο για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Όπως ξέρετε, για μας από τη Δύση, τους άλλους ε, που είμαστε σχετικά νέοι, για μας η Σλοβακία δεν είναι ουδέτερη χώρα. Εγώ όταν ήμουν 13 είχαμε την άνοιξη της Πράγας όπως τη λένε, αλλά ήταν και άνοιξη της Βρατισλάβα. Τότε είδαμε στη Σλοβακία και τις πρώτες κινητοποιήσεις. Και βλέπουμε με ιδιαίτερη προσοχή τη χώρα αυτή, με αγάπη. Υπάρχει ελπίδα που γεννιέται σε αυτή τη χώρα και οι Σλοβάκοι δεν θα πρέπει να πιστεύουν ότι δεν αγαπούν ε, οι άλλοι Ευρωπαίοι την ε, Σλοβακία, γιατί συμβαίνει ακριβώς ε, το αντίθετο, όπως και οι Σλοβάκοι αγαπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε. Υπάρχουν και διάφορα περιστατικά. Παραδείγματο χάρη, εξόριστη κυβέρνηση τη τότε Τσεχοσλοβακία μαζί με άλλε κυβερνήσει τη Κεντρική Ευρώπη είχε ε, καταρτήσει ένα προσχέδιο για την Ευρώπη που το έλεγε ε, σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι γνωστό αυτό το κείμενο. Στο τέλος του υπάρχει μια φράση που πάντοτε με εντυπωσίαζε και με συγκινούσε. Οι χώρε αυτέ τη κεντρική Ευρώπη με την εξόριστη κυβέρνηση έγραφαν μια τελευταία φράση που έλεγαν ότι μια μέρα Θέλουμε οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης να έρθουν μαζί μας για να οικοδομήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιστορία σας εμπόδισε να είστε εσείς που θα ε, δώσετε αυτό το όνομα, αλλά αφού η κέντρο Ευρωπαίοι ήταν αυτοί που πρώτοι οραματίστηκαν μια ειρηνική Ευρώπη, είναι δικό μας καθήκον να συνεχίσουμε το δικό σας έργο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστουμε Ζαν Κλόντ. Και τώρα να ξεκινήσουμε με τις παρεμβάσεις εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Πρώτος ο κύριος Γκονζάλες Πόντς, εκ μέρους του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Γιούγκερ για τα λόγια σας. Ευχαριστώ και τον Πρωθυπουργό, τον οποίο θέλω να καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί σα το όραμά σα για την Ευρώπη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Σα ευχαριστούμε και για τον τόνο σα και για τη γλώσσα σα. Και επίση, ε, αναφερθήκατε στη δολοφονία του Γιάνν Κούτσακ και τη συντρόφου του Βέβαια, δεν είναι αρκετή η μόνη αναφορά. Η ελευθεροτυπία είναι ένα από του σημαντικότερου πυλώνε τη δημοκρατία. Και όταν δολοφονείται ένα δημοσιογράφο, η τραγωδία αυτή πλήττει όλες τις δημοκρατίες. Ε, στη Μάλτα ακόμη κανείς δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη για την δολοφονία της Ντάφνη Καρουάνα, το οποίο μας λυπεί και το καταγγέλουμε. Στη Σλοβακία πέραν ε, τη παρέτηση ε, του ΦΥΚΟ, του δεν έγινε κάποια σημαντική πρόοδο. δεν έχει ολοκληρωθεί καν η έρευνα. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Ε, επίσης, Κάτι το οποίο μας ανησυχεί πολύ είναι η ρητορική ορισμένων αμελών του συνασπισμού σα ή ε, προεδρικών υποψηφίων που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ρητορική μίσο κατά της αντιπολίτευση, ρητορική μίσο κατά του τύπου. Εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε σχετικά. Είστε πραγματικά προσιλωμένος στον αγώνα κατά του εξτρεμισμού και της ρητορικής μίσους που κάποιοι αρκετά κοντά σας ε, χρησιμοποιούν. Έρχονται δύσκολοι καιροί για την Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν. Δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσει το Brexit. Ε, η Διατλαντική Συμμαχία επίσης ε, τίθεται από αφισβήτηση. Η ρωσική κυβέρνηση προσπαθεί να μας αποδυναμώσει, να μας διαιρέσει για να επικρατήσει. Υπάρχει μεγάλη μεταναστευτική κρίση, μια άνευ προηγουμένου κρίση με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι πραγματικότητες αυτές που πρέπει για να αντιμετωπιστούν να είμαστε πιο ενωμένοι. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι μα. Όταν είμαστε σε τέτοιε συνθήκε, ε, φαίνεται η δική σα κυβέρνηση να ζητά ε, μια διαφορετική προσέγγιση. Ε, άλλα λέτε εδώ. Και η κυβέρνησή σα, η χώρα σα κάνει τα αντίθετα. Ποια είναι η θέση σα πραγματικά η θέση σας ε, εκφράζεται σε αυτά που είπατε εδώ ή σε αυτά τα οποία πράττει η κυβέρνησή σα, στη Σλοβακία. Είστε ε, προσιλωμένο ε, στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. ανήκει η χώρα σας στο ΝΑΤΟ στο Βορτλαντικό Σύμφωνο. Είναι ερωτήσεις αυτές γιατί ε, μας ανησυχούν αυτά τα θέματα ε, και νομίζω ότι ε, σήμερα τα λόγια σας έρχονται σε αντίθεση με τα έργα της κυβέρνησής σας. Εμείς στο ΕΛΚΑ πολύ ξεκάθαρα ξέρουμε ότι την Ευρώπη πρέπει να την οικοδομήσουμε πάνω σε συγκεκριμένες δράσεις στην, πάνω στην βάση της κοινωνίας, όχι στη σελίτα. Η γεωργία ε, είναι ένα πρόβλημα η διαχείριση ε, όπως γίνεται σε συγκεκριμένες χώρες. Δεν μπορούμε την εθνική πολιτική να την βασίζουμε στην αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες, ε, σε ένα πολιτικό πόλεμο. Ο ευρωλαϊκισμός και ο εθνικός λαϊκισμός αλλά και ο ευρωλαϊκισμός είναι επικίνδυνες τάσεις. Υπάρχουν λογικές μάχες, κύριε Πρωθυπουργέ, που Μπορεί να μην γίνονται ε, σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά είναι ε, παρόλα αυτά σημαντική ιδεολογική πόλεμη για την Ευρώπη, ε, όπως αυτό που βλέπουμε να γίνεται με τη Βενεζουέλα για το Γουαϊδό. Ε, δεν τον έχετε ε, αναγνωρίσει. Άρα μπείτε, μπαίνετε στην τροχιά του Ιράν και της ε, Ρωσίας. Πόσο, κύριε Πελεγκρίνη, θα χρειαστεί για να σταθείτε στο πλευρό των ανθρώπων που πεινούν και δεν έχουν τρόφιμα, που είναι άρρωστοι και δεν έχουν φάρμακα. Άρα, ενότητα. Ενότητα από όλους, για όλους, ιδεαλισμός, επαφή με τους πολίτες μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά. Γιατί όλο και περισσότεροι πολίτες αποστρέφουν το βλέμμα τους ε, ε, και προσελκύονται από τα εξτρεμιστικά και λαϊκιστικά ε, κινήματα. Σίγουρα είναι μια τεράστια απειλή στο ευρωπαϊκό έδαφος ο εθνικολαϊκισμός. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή. Όλες οι άλλες υπάρχουν βέβαια και οι απειλές, αλλά αυτή διαβρώνει και διαβρώνει πολύ περισσότερο γιατί έρχεται από μέσα στο επόμενο κοινοβούλιο θα έχουμε λαϊκιστές, εθνικιστές, ε, θα έχουμε μια μεγάλη πολιτική ομάδα που θα παρτίζεται από τέτοιους πολιτικούς και εμείς ε, και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εσείς ως Συμβούλιο σύντομα έχετε ένα πολύ σημαντικό έργο να επιτελέσετε. Πρέπει να προτείνετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν πρόεδρο ε, και ελπίζω αυτό για την Κομισιόν. Ελπίζω να καταλήξουμε σε μια δέσμευση, να μην δεχθούμε υποψήφιο που ήταν υποψήφιο σε ευρωεκλογέ κατά το παρελθόν να μην ε, μας τον επιβάλλει κάποιος, αλλά να ψηφιστεί. Ε, στις 26 Μαΐου θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ιστορία που θα πρέπει να γίνει η οικοδόμησή του με συνεργασία. Πρέπει να ακουστούν όλες οι φωνές, μεγάλες και μικρές, όλες οι φωνές, διότι το μεγαλείο της Ευρώπης είναι ενότητά της. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, ήταν ε, λόγια έμπνευση ε, αυτά τα οποία ε, είπατε για την Ευρώπη, για τον ρόλο της Σλοβακίας, μια χώρα που είναι στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ δύση και Ανατολής, που είναι στο κέντρο της Ευρώπης, που όμως την ενώνει, ενώνει αυτές τις δύο πλευρές και ο Δούναβης. Ε, και πραγματικά είναι μια χώρα που έχει να επιδείξει ε, εκπληκτική πρόοδο ε, και η απόσχηση της Τσεχοσλοβακίας, η διαίρεση της Τσεχίας και Σλοβακία έγινε με πάρα πολύ ομαλό και επιτυχημένο τρόπο. Επίσης για το ευρώ πλήρωσε τα κριτήρια η Σλοβακία και αυτό οδήγησε σε οικονομική ανάκαμψη. Είναι πάρα πολύ θετικά όλα τα δείγματα, είναι σε καλό δρόμο η Σλοβακία έγινε ένας παράγοντας πρόοδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως υπάρχουν και κάποιες σκιές ακόμη. Ε, υπάρχει ε, επιρροή από τη μαφία, υπάρχει διαφθορά σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η ερευνητική δημοσιογραφία δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα ε, με τη δολοφονία ε, του ε, Κούτσιακ και πραγματικά αυτό συντάραξε, συγκλώνησε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και σίγουρα νιώσατε τις πολιτικές συνέπειες και στη χώρα σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συγκροτήσει αυτή η ομάδα κράτους δικαίου στο πλαίσιο Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και στην επόμενη είναι ολομέλεια. Ε, θα ψηφίσουμε μια σχετική έκθεση. Είναι σε πολύ σημαντικούς τομείς θετικός απολογισμός ε, ε, της χώρας σας. Υπάρχουν σημαντικοί στόχοι οι οποίοι έχουν επιτευχθεί, Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκή Προστέμενη Αξία. Υπάρχουν όμως αμφιβολίες για το κατά πόσον έχετε προωθήσει επαρκώ ε, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την ελευθεροτυπία και έχετε ε, συναγάγει ε, τα απαραίτητα συμπεράσματα. Εμείς θα σα στηρίξουμε να έχετε έναν μηχανισμό κράτος δικαίου που θα είναι ανεξάρτητο από τραγικά συμβάντα σαν αυτά που βιώσαμε κατά το παρελθόν. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας σας, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ασφάλεια των πολιτών. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να επιβάλλουμε κάτι. Θέλουμε να, γίνονται, να εφαρμόζονται οι κοινοί ε, κανόνες ε, ε, που μας ενώνουν Δύση και Ανατολή. Μίλησε ο κύριος ε, Γιούνκερ για τους δύο πνεύμονες ε, της Ευρώπης. Πραγματικά πρέπει να δούμε με κριτικό πνεύμα τη Δυτική Ευρώπη και υπάρχουν προβλήματα σίγουρα δεν μπορούμε πάρα πολύ ε, ε μα, κέρδη να έχουμε, ε, παραδείγματο χάρη με πολύ ψηλού ε, συντελεστέ. Επίση, φυγή εγκεφάλων ε, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τι ανισορροπίε και θα σα στηρίξουμε σε αυτέ σα τι προσπάθειε. Παραδείγματο χάρη. Ε, η το επίδομα ε, για την ανεργία. Είναι κάτι που πρέπει να προχωρήσει και άλλες πρωτοβουλίες για να μην καταρρεύσει, για να μην διαλυθεί η Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να κοιτάμε βραχυπρόθεσμα μόνο ωφέλη. Επίσης, επίτευξη των στόχων του κλίματος. Δεν θα πρέπει αυτό να το καθυστερούμε και να το αναβάλουμε πάοριστον. Γιατί είναι θέματα που μας αφορούν όλους και στη Δύση και στην Ανατολή. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, με δικαιοσύνη ε, κοινωνική, ε, με ισότητα. Και δεν είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας ε, και κυριαρχίας. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, προσανατολισμένοι στο μέλλον για να προχωρήσουμε. Έτσι μόνο θα αναπτυχθούμε, αν μπορούμε να βρούμε κοινέ λύσεις. Θέλουμε λοιπόν κατώτατο μισθό, ίση αμοιβή για την ίδια εργασία, ψηφιακή Επανάσταση και τα λοιπά Η κοινωνική Ευρώπη είναι η καλύτερη εργαλειοθήκη για μια ε, καλύτερη Ευρώπη. Έχετε ήδη κάνει σημαντικά πράγματα εσείς στη Σλοβακία, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να προσφέρετε ακόμα ένα μεγαλύτερο λιθαράκι. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, η κυρία Ζετνάνσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, πριν από 20 χρόνια είχαμε τη διεύρυνση, την πρώτη διεύρυνση του ΝΑΤΟ μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Σλοβακία δεν πήρε τότε μέρος. Όμως στη συνέχεια συμμετείχαμε και εμείς, όχι μόνο στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, αλλά αργότερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς όμως όλα αυτά έχουν ε, τεθεί ένα αμφιβόλο όχι μόνο από εξτρεμιστικές κυβερνήσεις αλλά και από το δικό μας το κυβερνητικό συνασπισμό. Το να ε, σμικρίνουμε το, τη σημασία της ε, στρατηγικής μας συμμαχίας προς συμφέρον της Ρωσίας είναι κάτι που βλάπτει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σλοβακία. Δεν μπορούμε να μην είμαστε αξιόπιστοι ως εταίρος για τους συμμάχους μας. Πρέπει να είμαστε και να έχουμε συνοχή στην πολιτική μας αλλά και για τα εσωτερικά της Τσεχοσλοβακία. Δεν μπορούμε διαρκώ να υποδαβλίζουμε φόβου στον κόσμο για να αποσπάμε περισσότερε ψήφου. Ε, πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι εύκολο να εκμεταλλευτεί κανεί τα αρνητικά συναισθήματα, όμω αν ξεφύγουν από τον έλεγχό του μπορεί να γίνουν και καταστροφικά. Τώρα λοιπόν πρέπει να